των Ο κύριο Μάρκο Τσάνι έφυγε από την ομάδα EFTD και προσχώρησε στην ομάδα ENF από τις 11 Ιανουαρίου. Ο κύριος Μάρκο Αφρόντε έφυγε από την ομάδα EFTD και προσχώρησε στην ομάδα των Πρασίνων από τις 11 Ιανουαρίου.